να ε, συνεχίσω να προεδρεύω κατά τη διάρκεια των ε, επεξηγήσεων ψήφου. Περιμέναμε λίγο για να παραμείνουν όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν το λόγο και να ακούσουν και οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν. Ε, θυμίζω σε εκείνους που έχουν παραμείνει στην αίθουσα και θέλουν να μιλήσουν ότι εδώ έχουμε επεξηγήσει ψήφου και παρακαλούνται οι ιδιωτικές συνομιλίες εκτός της αιθούσης να συνεχιστούν. Λοιπόν, Έχουμε τώρα την έκθεση του κυρίου Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε και του κυρίου Μπούλμαν με θέμα την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Πέντε συνάδελφοι παρακάλεσαν να τους δοθεί ο λόγος για επεξήγηση ψήφου. Πρώτος, ο κύριος Μόμτσιλ Νέκοφ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων ήδη ε, λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Όμω βλέπουμε να υπάρχει μια σαφή διάκριση μεταξύ Ανατολή και Δύση. Τον Ιούλιο του 2016 η μεγαλύτερη στήριξη προς τα κράτη-μέλη είχε πάει στα δυτικά κρατημέλη με 91% του συνόλου του χαρτοφυλακίου του, ενώ πολύ μικρά ποσά στα υπόλοιπα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει υποστηρίξει έργα τα οποία ε, αφήνουν πολλές αμφιβολίες σε σχέση με τα κριτήρια ρεσιμότητας. Εδώ και χρόνια ακούμε από το βουλγαρικό κόμμα ΓΚΕΡΠ ότι αυτό το ταμείο θα μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερες διασυνδέσεις στη χώρα, αλλά μέχρι τώρα έχουμε μόνο υποσχέσεις. Ελπίζω ότι αυτό το πρόγραμμα με την αναθεώρησή του θα ε, θέσει τις σωστές προτεραιότητες και δεν θα παραμείνει μόνο στα λόγια των εκστρατιών. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί Γερμανοί συνάδελφοι, πολύ ενδιαφέροντα σίγουρα αυτά που λέτε, αλλά δεν μας αφορούν εμάς. Η κυρία Νταμάτο, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. μπορούμε να λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων είναι σαν καλό κρασί, αλλά θα μεθύσουμε αν συνεχίσουμε να κοιτάμε μόνο του αριθμού του. Πρέπει λοιπόν να ε, ξεφύγουμε από την αφήγηση για ένα ε, πρόγραμμα επενδύσεων που θα στηρίζει τις μικρομεσαίες, την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Έχουν υποτιμηθεί οι δείκτε, δεν υπάρχουν πληροφορίε για τι θέσει εργασία που έχουν δημιουργηθεί, για τη λειτουργία των διαδικασιών και του αριθμού που αποκρύπτονται. Ακόμη και το ελεγκτικό συνέδριο είπε ξεκάθαρο ότι έχει πολύ περιορισμένο αντίκτυπο το ΕΦΣΥ. υπάρχουν έργα που έχουν σχέση με ορεικτά καύσιμα όπως το, το πετρέλαιο και το αέριο, το φυσικό αέριο. Τίποτα δεν γίνεται για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για τις ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας ε, και ούτε αναλαμβάνονται έργα υψηλού κινδύνου. Εξυπηρετεί τις τράπεζες το ε, πρόγραμμα αυτό και μπορεί να γίνει ρολακική βόμβα για την πραγματική οικονομία. Γι' αυτό το λόγο το καταψηφίσαμε. Ευχαριστώ. Μιλήσατε περισσότερο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Και τώρα ο κύριος Χάναν. Ευχαριστώ. Το χρήμα είναι όλο το θέμα, έτσι. Πόσες φορές δεν έχουμε περάσει στην αίθουσα αυτή οι συζητήσεις για να μιλάμε για μεταφορέ ε, ποσών. Και δεν σκεφτόμαστε τι αντίκτυπο θα υπάρχει για τα άτομα, τους πολίτες, ε, αυτούς που θέλουν να εργαστούν, τους εργολάβους, ε, τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Βρυξελών και θέλουν να κερδίσουν τη ζωή τους. Έχουμε βρει καινούργια γλώσσα για να ε, χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να κάνουμε το χρήμα να κυκλοφορεί και να περιγράφουμε αυτή την κίνηση του, όπως το grid, το δίκτυο, που... Αλλά όλα αυτά είναι απλή πλεονεξία. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εάν ψηφίσετε πολιτικούς που υπόσχονται να σας τα χρήματα άλλων, μην παραπονιέστε όταν σας παίρνουν τα λεφτά πίσω για να τα ε, χρησιμοποιήσουν για τον εαυτό τους. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ανδρέας Μαμίκινς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενθύσεων ε, είναι προς όφελος εκείνων των χωρών που δεν έχουν προβλήματα επενδυτικά ούτε γεωγραφική κατανομή. Ε, τώρα συνεχίζει ο ανταγωνισμός και για τη λετωνική οικονομία ε, έχουμε κάποια αποτελέσματα, αλλά με τεράστια δημογραφική αλλαγή. Πολλοί έχουν φύγει από τη χώρα γιατί έχουν κουραστεί να περιμένουν να φτάσει σε επίπεδα Δυτικής Ευρώπης η Λετωνία. Ε, προσπαθούν, ε, προτιμούν να φύγουν με τις οικογένειές τους προς τη Δύση και δεν υπάρχει προοπτική για εκείνους που παραμένουν. Είναι μια χώρα όμορφη αλλά άδεια με μια, ένα μικρό πληθυσμό φτωχό και ηλικιωμένο. Ε, η Λετωνία χρειάζεται επενδύσει από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και η κατανομή θα πρέπει να γίνεται αδιακρίτω. Υποστηρίζω την έκθεση και ιδιαίτερα την ιδέα να δοθεί τεχνική βοήθεια στι χώρες εκείνες και τι περιφέρειες που έχουν αποφεληθεί λιγότερο μέχρι σήμερα από το ΕΦΣΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στα λετωνικά λέει ο Πρόεδρο. Ε, η κυρία Άννα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι εγώ υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για έναν τρόπο προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης έργων για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία. Είναι πολύ καλές οι προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το νέο αυτό εργαλείο και πώς να βελτιωθεί η επικοινωνία με τους πολίτες και τον επιχειρηματικό κόσμο. Το επενδυτικό κλίμα και η βελτίωσή του όμως δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τις δημόσιες επενδύσεις αλλά και προσέγγιση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Dante για την ε, συνεργατική οικονομία. Πρώτη επεξήγηση ψήφου θα γίνει από τον κύριο Τίμπορ Σάνι, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Σάνι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση Dante για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Συνεργατική Οικονομία και χαιρετίζω την ιδέα γιατί ενισχύει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει θετικά και τα εργασιακά δικαιώματα, όπως αναφέρεται στο κείμενο. Επίσης, υπερψήφισα γιατί δεν ξεχνάμε στην έκθεση και τις αγροτικές περιοχές. Η συνεργατική οικονομία δίνει μεγάλες ευκαιρίες στις αγροτικές περιοχές και στις μειονεκτούσες περιοχές. Γι' αυτό και υπερψήφισα. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Άντρης Μαμίκινς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνεργατική οικονομία δημιουργεί νέε ευκαιρίε για τι κοινωνίε μα και είναι και σημαντική συνεισφορά για τη δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βασική πρόκληση είναι να βρούμε το σωστό ορισμό. Τι εστί συνεργατική οικονομία η απάντηση ε, έτσι θα βοηθήσει για ε, καλύτερη προστασία των καταναλωτών, ε, εργασιακές σχέσεις κλπ. Η συνεργατική οικονομία επιτρέπει στους ανθρώπους να εργάζονται με ευελιξία και να μπορούν να δραστηριοποιούνται οικονομικά, ενώ πιο παραδοσιακή, εκεί που εκεί που πιο παραδοσιακέ μορφέ εργασία δεν προσφέρονται. Χρειάζεται προσοχή όμω, γιατί οι πλατφόρμες και η τεχνολογία χρησιμοποιούνται πολλέ φορέ για να παρακάμψουν ε, την εργατική νομοθεσία ε, και τι συνθήκε εργασία και τη φορολογία. Γι' αυτό βλέπουμε μια κούρσα προ τα κάτω που μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά. Ε, η συγκεκριμένη έκθεση είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενη μιλήτρια, η κυρία Λούση Άντερσον. Όχι, η κυρία Ζαμπόσκα λέει ο πρόεδρος. Α, ζητώ συγγνώμη. Εγώ φταίω. Ε, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Η κυρία Λούση Άντερσον εννοούσα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η συνεργατική οικονομία σε τομείς όπως οι μεταφορές μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και να δημιουργήσει ποιοτικέ θέσει εργασία. Πρέπει όμω να ρυθμιστεί με υπεύθυνο τρόπο για να προστατεύσουμε τι προσδοκίε των εργαζομένων και πολιτών που εμπλέκονται σε αυτά τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα επίση. Είναι ύψιστη τη σημασία να βεβαιωθούμε ότι η φορολογία και άλλε προτεραιότητε τη δημόσια και κρατική πολιτική ρυθμίζονται σωστά από τα μέτρα αυτά που προβλέπονται για τη συνεργατική οικονομία. Το κείμενο αυτή τη έκθεση αντικατοπτρίζει αυτέ τι ανησυχίε και με μεγάλη χαρά το υπερψήφισα. Ευχαριστούμε. Κύριε Άντερσον, με συγχωρείτε και πάλι που σας παρέλειψα. Η κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα την πρόταση αυτή για τη συνεργατική οικονομία, αν και είχα κάποιες επιφυλάξεις αρχικά. Γιατί νόμιζα ότι δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στη συνεργατική οικονομία και την οικονομία της αγοράς. Χαίρομαι που εκθέσεις πρωτοβουλίας όπως αυτή διευρύνουν τον ορίζοντα της σκέψης μου και μου δίνουν τη δυνατότητα να έχω μια νέα ματιά ε, απέναντι σε γνωστά φαινόμενα όπως είναι η κατανομή της εργασίας, ο επιμερισμός, η συνεργασία στην ανταλλαγή και ε, ε, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Θα περάσει όμως μάλλον πολλή χρόνος μέχρι να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με τη συνεργατική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ζαμπόρσκα. Περνάμε στην επόμενη έκθεση των Βιρκούνεν και Ζουβά για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ο κύριος Μόμτσιλ Νέκοφ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι η ψηφιακή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά κατακαιρματισμένη, κάτι που μειώνει την ανταγωνιστικότητά της παγκοσμίω. Επίσης υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου, κάτι που δημιουργεί δυσκολίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εξάλλου η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη επικοινωνικών πλατφορμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να φτάσουν και να διεισδύσουν στην παγκόσμια αγορά. Και με αυτή την ε, επιγραμμική πρόσβαση των νεοφυών ε, νεοσύστατων εταιριών κάνουμε οικονομία και στις επενδύσεις. Μιλούμε άλλωστε και για το δίκτυο 5G. Στις περισσότερες όμως αγροτικές περιοχές της Βουλγαρίας δεν έχουμε ούτε καν 3G, για να μην πω 4G. Γι' αυτό λοιπόν τάχθηκα υπέρ της έκθεσης. Μπλαγκανταριά. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Στίβορ Σάνι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η έκθεση αναφέρεται στις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις της αφορά την, τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας 5G και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τις σχετικές υποδομές και να κάνει τις αντίστοιχες επενδύσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ε, πρόσβαση και στο βριζονικό ίντερνετ υψηλή ταχύτητα ε, και στι αγροτικέ περιοχέ, και εν καιρό και στο δίκτυο 5G. Θα πρέπει να μειώσουμε έτσι τι ανισότητε μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι δεμοί θα υστερούν όλο και περισσότερο εξαιτία έλλειψη πρόσβαση σε αγροτικέ περιοχέ και δεν θα μπορούν να πτήσουν τι ψηφιακέ του δεξιότητε, ε, οι κάτοικοι τους. με την πρόταση αυτή θα βοηθήσουμε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις ε, να κάνουμε κάτι και για την ε, αποφυγή της εξάπλωσης χαλκευμένων ειδήσεων fake news και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σον Κέλλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή και ευχαριστώ τους ε, εισηγητές Φερκούνεν και Ζουβέν για τη δουλειά του και τη δημιουργία, την προσπάθεια δημιουργία πλέον ευκαιριών για τι προγραμματικέ πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά. Χρειάζονται ε, προσπάθειε καινοτομία εδώ, νέες ευκαιρίε και αντιμετώπιση των προκλήσεων στο σχετικό τομέα. Η έκθεση σωστά εξετάζει από τη σκοπιά της συνεργατικής οικονομίας τις δυνατότητες ε, μεταφοράς δεδομένων στις επιγραμμικές πλατφόρμες καθώς και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την ε, οικοδόμηση τέτοιας ενιαίας ψηφικής αγοράς για το μέλλον. Γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση αυτή και εύχομαι όσο δυνατόν συντομότερα μικρομεσαίε επιχειρήσει και οι πολίτε να μπορέσουν να υποφεληθούν από τα όσα προβλέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. επόμενες επεξηγήσεις ψήφου από το ψήφισμα για την ανθρωπιστική κατάσταση της Ιεμένης. Ο πρώτος είναι κανονικά ο κύριος Φαρία, απουσιάζει όμως, δεν τον βλέπω στην αίθουσα, οπότε περνάμε στον κύριο Αντρέης Μαμίκινς. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σύγκριση στην Ιεμένη δεν κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωση στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε το κλασικό πρόβλημα επιλεκτική τυφλότητα στην Ευρώπη. Ε, γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την Ιεμένη. Αλλά ένα πρόβλημα υπάρχει στην Ευρώπη μόνο όταν το βλέπεις στην τηλεόραση και στα social media και είναι συναισθηματικά φορτισμένο και δημιουργεί εντυπώσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει, δεν το γνωρίζουν. Άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να λυθεί αυτή η αιματηρή σύραξη. Πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν είναι ειλικρινείς ε, Ορισμένες πολιτικές ελίτ ε, ενδιαφέρονται ε, να πουλάνε όπλα στη Σαουδική Αραβία και ως γνωστό τα λεφτά δεν έχουν οσμή. Πραγματικά ε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρεσκόμαστε έτσι να κρίνουμε και να επικρίνουμε τους άλλους, αλλά δεν κάνουμε αυτοκριτική. Ιδιαίτερα ε, ε, η Γκούι και οι ε, Πράσινοι νομίζω είχαν την κατάλληλη στάση στο ψήφισμα. Ευχαριστώ. Περνάμε στην τελευταία φάση των επεξηγήσεων. Έχουμε καταρχήν το ψήφισμα για το καθεστώς και την χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων. Έχουμε εδώ τέσσερις ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Τιμποσάνη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα ε, την έκθεση αυτή, το ψήφισμα για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε τον κανονισμό 1041 και να επιτρέψουμε καλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν κάποιε αδυναμίε. Θα πρέπει να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προτείνει την αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μιχαέλα Σόιντροβα για ένα λεπτό από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. υπερψήφισα το, το ψήφισμα αυτό για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, διότι η δημοκρατία χρειάζεται δημοκράτες, καθώς και ελεύθερους υπεύθυνους πολίτες. Νομίζω ότι το τωρινό σύστημα επιτρέπει Δυστυχώ να ανθούν τα αντιευρωπαϊκά κόμματα. Γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδεί τον ε, ισχύοντα κανονισμό. Ε, στήριξα ε, όλος ιδιαίτερος το στοιχείο της διαφάνειας. Διαφάνεια που θα είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί, καθώς και ο περιορισμός των αριθμών, του αριθμού των βουλευτών, που θα πρέπει να είναι γνωστές οι, το πιο ποιο ακόμα ε, ανήκουν. Και περνάμε στους τρεις τελευταίους ομιλητές. Είναι όλοι από τη Σλοβακία. Κυρία Ζάμπορσκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα, πρέπει να σας πω ότι ε, το Κοινοβούλιο απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Συμφωνώ ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές ε, στη χρηματοδότηση, αλλά επίσης κατανοώ και τις ανησυχίες και τους φόβους των μικρών πολιτικών κομμάτων ε, ε, γιατί οι συγκεκριμένες αλλαγές μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες για αυτούς. Άρα είμαι πεπισμένη ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να προχωρούν με σύνεση και προφύλαξη προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, να την αξιολογήσουμε ε, και να δραστηριοποιηθούμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το τελικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν θα επιδέχεται αλλαγές και βελτιώσεις. Επίσης επιμένω στο μέλλον να αλλάξουμε τους κανόνες ε, έτσι ώστε οι αλλαγές να ισχύουν από την επόμενη ε, θητεία. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντική η παρέμβασή σας και σας ευχαριστούμε για την αιτιολόγηση. Ο κύριος Μπράνισλαβ Σκρίπεκ για ένα λεπτό είναι και ο τελευταίος μας ομιλητής στις αιτιολογίες ψήφου. Ευχαριστώ. Κάθε τρεις και λίγο προσπαθούμε να αλλάξουμε τους κανόνες για τα ευρωπαϊκά κόμματα. Κάθε φορά έχουμε συζήτηση και πολλή δουλειά, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι καλό για μια σταθερή δημοκρατία όπως είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα ε, η πρόταση αυτή δεν μας βοηθά με τον αριθμό που προτείνουμε, ε, γιατί δεν ενισχύει το διάλογο Ευρωπαίων πολιτών και Ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών. Δίνει την εντύπωση ότι πρέπει να είναι κανεί μέσα στην υποφόλυγα των Βρυξελών για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Και αν θέλουμε τρει ως πέντε βουλευτές να δημιουργήσουμε ακόμα, ουσιαστικά θα κλείσουμε την πόρτα για οποιαδήποτε πρωτοβουλία από τη βάση. Τέτοιου είδου πρωτοβουλίε όμω χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι όλα τα μικρά και νέα κόμματα κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα έτσι δεν θα σταματήσουμε τι ακροδεξιέ ε, δυνάμει, αλλά είναι αντιδημοκρατική η πρόταση και ει βάρο όλων των μελλοντικών κομμάτων. Δεν είναι αυτό το κατάλληλο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στου Ευρωπαίου πολίτε μα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σκρίπεκ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που έμειναν στην αίθουσα. Είναι οι πιο αθεκτική πραγματικά. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, ε, τους υπαλλήλους μας από τη διοίκηση. Θα διακόψουμε για το μεσημέρι. Σας εύχομαι καλή όρεξη και διακόπτουμε μέχρι τις 3.